Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη συνεδρίασης. Έχετε την ημερήσια διάταξη, το σχέδιο, μπορούμε να την εγκρίνουμε όσοι έχει υποβληθεί, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 21ης και 22ης Ιανουαρίου και αν δεν διαφωνείτε εγκρίνονται και τα πρακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τρίτον, ενημέρωση από τον τριμερή διάλογο σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος του Λιμένα. Είναι δική μου έκθεση. Σύμφωνα με το άρθρο 70 του κανονισμού θα ήθελα να σας ενημερώσω για τον πρώτο τριμερή διάλογο που είχαμε με την Ελλαδική Προεδρία για το κράτος Λιμένα. Έλαβε χώρα εδώ στο Κοινοβούλιο στις 30 Ιανουαρίου Παρουσία της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου που απαρτίζεται από τον υποφαινόμενο εισηγητή και όλους τους σκιώδεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από τον κύριο Καραμίτσο. Θα ήθελα να σας ε, θυμίσω ότι αυτή η αναθεώρηση έχει να κάνει με την ενσωμάτωση ε, της ε, Σύμβασης για την Ναυτική Εργασία του 2006 ε, στην Οδηγία για τον έλεγχο του κράτους λιμένα. Όπως πολλές διεθνείς συμβάσεις και αυτή ε, υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να κάνουν επιθεωρήσεις στα λιμάνια. Και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ φέτος τον Αύγουστο αυτή η Σύμβαση για την Ναυτική Εργασία. Οπότε καλό θα ήταν να τεθεί σε ισχύ και σε εφαρμογή και να υλοποιείται το συντομότερο δυνατόν. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του τριμερούς διαλόγου έγινε εκτατική συζήτηση για δύο σημεία που είναι από τα πιο επίμαχα, ε, το θέμα της ε, ε, μη κύρωσης και της μη οπισθοχώρησης στην προκείμενη κατάσταση. Οι θέσεις μας με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που έχουν πάρα πολύ για τη μη κύρωση Ε, ε, Ευρωπαϊκή, το Συμβούλιο δεν συμφωνεί ε, να συμμετέχουν κράτη που δεν έχουν κυρώσει μία ή περισσότερες συμβάσεις και εμείς συμφωνούμε θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού γενικότερα στην αυτιλία. Ε, σε ό,τι αφορά τη ρήτρα ε, για τη μη ε, οπισθοχώρηση, οπισθοδρόμηση, φρονούμε ότι υπάρχουν ισχυρές εγγύσεις στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην θεωρημένη οδηγία για το έχω του κράτους λιμένα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει οπισθοδρόμηση σε σχέση με τα εργατικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Τελικά η Ιρλανδική Προεδρία ε, έκανε μια συμβαστική πρόταση που δεν τη δεχτήκαμε. Ε, θα γίνουν και άλλες συζητήσεις στις ερχόμενες εβδομάδες για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την υπόθεση και για αυτό το σημείο. Και πολλά άλλα σημεία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, όπως και άλλες συμβαστικές προτάσεις που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία. Χαιρετίζω το συμβιβασμό που προτάθηκε για την προστασία της ε, ε, εμπιστευτικότητας του απορρίτου των καταγγελιών ορισμένων ναυτικών. Στις 27 Φεβρουαρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση τριμερούς διαλόγου και ελπίζουμε να συνεχίσουμε εκεί τις συζητήσεις με την Ελλαδική Προεδρία. Αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα ότι θα καταλήξουμε σε αυτή τη συνεδρίαση. Παρ' όλα αυτά ελπίζω να κάνουμε κάποια πρόοδο. Αυτά είχα να σας αναφέρω από τη συνεδρίαση αυτή του τριμερούς διαλόγου για το έλεγχο κράτους λιμένα. Έχει κανείς ερωτήσεις ή σχόλια να κάνει. Εάν όχι, να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση. Ε, προσωρινή παρέκκληση από την οδηγία και τα λοιπά Είναι του κυρίου Γκρός για την ενέργεια κυκλοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και παρόλα αυτά προσπαθήσαμε και να επιτύχουμε συμβιβασμό και βεβαίως την έκθεση και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν δραστήρια. Γενικά πιστεύω ότι αυτή αυτή η θέση που διαγράφεται ε, στοχεύει στο να σταματήσει το ρολόι για ένα χρόνο. Και αυτό θα, είναι, θα δώσει ένα μήνυμα έτσι ώστε τα κονδύλια τα οποία συλλέγονται από το σύστημα εμπορίας αερίων θερμοκηπίου ε, να παγιωθεί διότι ξέρουμε ότι πολλές φορές ανακύπτει το ζήτημα εκτός Ευρώπης μας ρωτάνε τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια, τι γίνεται με αυτά τα χρήματα, πώς διατίθενται, δεν μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Στα πλαίσια λοιπόν του συμβιβασμού και στη συζήτηση που κάναμε, η ε, ιδέα, η ε, ε, ιδέα τέθηκε η ιδέα να αυξήσουμε αυτό το, αυτή την αναστολή πάνω από ένα χρόνο, αλλά τελικά καταλήξαμε στο να αναστείλουμε για ένα χρόνο έως ότου συνεδριάσει το Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, του ΔΟΠΑ, ΙΚΑΟ εάν καταλήξουν τότε θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση που είπαμε εάν δεν καταλήξουν προς το δικό μας στόχο, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια ε, εκ νέου συζήτηση, δεδομένου ότι το, εάν δεν καταλήξουν θα αποδυναμωθούν και, αποδυναμωθούν και τα επιχειρήματά μας. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Θα δούμε τι θα προκύψει. Θα αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα της Συνόδου με την Κομισιόν και θα διευκρινίσουμε, θα τονίσουμε ότι θέλουμε και στο μέλλον να αποφύγουμε σαφώς τρευλώσεις του ανταγωνισμού. Ε, γι' αυτό ε, πρέπει να φροντίσουμε να συζητηθεί και το θέμα το ένδο ευρωπαϊκών πτήσεων, όχι να αναστείλουμε τα πάντα για ένα χρόνο και μετά να κάνουμε την αξιολόγηση. Ε, ναι, λοιπόν, ένα χρόνο να αναστείλουμε, να κάνουμε την αξιολόγηση μετά από το χρόνο αυτό και μετά να δούμε αν τυχόν έχει προκύψει κάποιο θέμα στρέβλωσης του ανταγωνισμού και να αξιολογήσουμε περαιτέρω την όλη κατάσταση. Αυτά αναμένουμε, αυτά συζητήσαμε, αναμένουμε τη θέση του ΙΚΑΟ. Υπάρχουν ορισμένοι που είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτή την αναστολή, άλλοι είναι πιο αισιόδοξοι. Εν πάση περιπτώσει, τηρήσαμε μια αντικειμενική στάση και ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συνεργάστηκαν ε, επικοδομητικά μαζί μου. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Ελχαντράου, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή εξαιρετική εργασία του, όσο και η ταχύτητά του, πρέπει να σας πω. Με αποτέλεσμα κάτι που ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε κι εμείς ως πολιτική ομάδα. Τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα συμφωνήσουμε να σταματήσουμε το για ένα χρόνο για μια προσωπική παρέκκληση δηλαδή για ένα έτος από την οδηγία αυτή. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνουμε γιατί ε, κάνουμε και ένα άνοιγμα προς τον ΙΚΑΟ έτσι για να καταλήξουμε παγκοσμίω σε μια συμφωνία και να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία ε, όλοι έτσι ώστε να καταπολεμούμε ε, την κλιματική αλλαγή και από πλευρά μεταφορών. Αλλά αυτή η προσωρινή παρέκκληση ε, δημιουργεί και μία πίεση, διότι κανείς ούτε εδώ στην Ευρώπη ούτε εκτός Ευρώπης έχει ε, πλεονέκτημα από μία πραγματική σύγκρουση. Βεβαίως θα πρέπει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να αξιολογήσουμε κατά πόσο μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα, αλλά δεν είναι του παρόντος αυτό, θα το δούμε το φθινόπωρο. Ένα σημείο μόνο, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να ε, τονίσω και να ζητήσω από τον εισηγητή να επιχειρηματολογήσει ή να επανεξετάσει ε, θέσεις του στις τροπολογίες 22 και 13 για την Ελβετία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρείται ότι υπόκειται στην νομοθεσία και η Ελβετία λόγω της συμμετοχής στο ΕΟΧ αλλά Ξέρετε, δεν είναι μια κοινή, μια τυχαία τρίτη χώρα. Δεσμεύεται και συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία με μια σειρά συμφωνιών και στις μεταφορές. Εγώ αγαπώ πολύ και συμπαθώ τους Ελβετούς ε, ε, φίλους. Καμιά φορά πολλές, ε, πρέπει να πω και περισσότερα από ορισμένου άλλους κράτη-μέλη. Αλλά Δεν μπορεί να εξαιρείται η Ελβετία και να μην υπόκειται στις ίδιες διατάξεις εταιρείες με τις δικές μας ε, πολιτικές εταιρείες. Ευχαριστώ, κυρία Μάισνερ. Yeah, Ευχαριστώ. Είχαμε συμφωνήσει τουλάχιστον να υπάρχει οπωσδήποτε αυτό το σύστημα εμπορίας αερίων στην Ευρώπη και γι' αυτό υπήρχε, παρουσιάστηκε και αυτή η πρόταση στο τραπέζι. Ήδη πολλά έχουν ελεγχθεί από τους προλαλήσαντες. Τώρα για να αρχίσουμε από το τέλος, στην Ελβετία υπάρχει ένα αίτημα να εξαιρεθεί η Ελβετία και το θέμα είναι είχε συμφωνηθεί η εξαίρεση τώρα μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε ο, κύριος, ο συνάδελφος κύριος Ελκαντρού είχε πει ότι είναι στην ε, Ευρώπη η Ελβετία και ότι θα μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε το θέμα είναι ότι έχει γενικά συμφωνήσει για το σύστημα εμπορίας η Ελβετία Ελπίζω να συμφωνήσουμε όμως, και αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα, σε διεθνές επίπεδο για το θέμα αυτό, διότι την περασμένη εβδομάδα οι Ηνωμένε Πολιτείε έδειξαν ότι δεν αναμένουν ε, λύση ε, στη Σύνοδο φέτος. Οπότε τίθεται το ερώτημα για μένα, εάν δεν υπάρξει ε, διεθνής λύση, πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε την εισαγωγή του συστήματος εμπορίας στην Ευρώπη, χωρίς να δημιουργήσουμε αρνητικές διακρίσεις έναντι των των ε, αεροπορικών εταιριών. Και γι' αυτό είχα, παραδείγματο χάρη με άλλου συναδέλφου, προτείνει να καλυφθούν, να εξαιρεθούν και οι εσωτερικέ ε, ευρωπαϊκέ γραμμέ ε, για να μην αποδυναμωθεί ο διεθνή ανταγωνισμό. Διότι διαφορετικά θα μπορούσαν οι αεροπορικές εταιρείες να προσγειώνονται και να χρησιμοποιούν αεροδρόμια εκτός Ευρώπης και όχι ενδοευρωπαϊκά, ενδοκοινοτικά ε, πιστεύω όμως ότι θα πρέπει οι εσωτερικές γραμμές, οι εσωτερικές πτήσεις να περιληφθούν. Πιστεύω ότι αυτό από απόψε ως αρχής είναι σωστό δηλαδή. Αλλά λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού, δεν θέλουμε κανέναν τρόπο να αποδυναμωθούν οι δικές μας εταιρείε, αεροπορικές εταιρείε. Τώρα το μορατόριο με αυτό θα αρχίσει μέχρι 1η ε, Μαΐου. Συνήθως η αξιολόγηση ε, γίνεται το φθινόπωρο. Τώρα θα γίνει τον Απρίλιο και να πούμε δηλαδή ε, το, το έτος αυτό να λήξει το τέλος του 2013. Τέλος του 2013 και με την προϋπόθεση ότι δεν θα επιτευχθεί διεθνής λύση. Με αυτό το, την αντίληψη πρέπει να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Κύριος Κράμορ, ευχαριστώ πολύ και ξέρω με της κυρίας Λίχτεμπεργκερ, ε, ε, τον εισηγητή, με την Ελβετία να δούμε τι θα γίνει. είναι πρόθυμοι να μας ακολουθήσουν, να τους κάνουμε την προσφορά. Αν την αρνηθούν, ε, δεν μπορούμε και να τους αναγκάσουμε. Ε, συμβιβασμοί μας βρίσκουν σύμφωνους και τους υποστηρίζουμε και κυρίως έχει ξεκαθαριστεί ότι αν δεν αλλάξει τίποτα στον ΙΚΑΟ και τεθεί σε ισχύ, είναι ένα απαραίτητο, ε, ε, και βέβαια ε, τι να κάνουμε, ε, θα πρέπει να πληρώσουμε και το τίμημα. Αν επιβάλλουμε ένα κόστος και ένα τέλος υπέπτυσης, μας λένε ότι δεν θα έρθει κανένας. Μα το κάνουν οι Ρώσοι για τη Σιβηρία και βγάζουν ένα σωρό λεφτά. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς. Ε, εντάξει, εμεί θέλουμε να έχουμε δίκαιο ανταγωνισμό και θεμητό στις αεροπορικέ εταιρείε, αλλά έχω ακούσει και από πολλούς ότι κυρίως ε, οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι διαφωνούν οι Ρώσοι είναι κατά διότι ε, αν γίνει κάτι τέτοιο για την αεροπορία θα μετατεθεί και στην αυσιπλοεία. Γι' αυτό θέλουν να το πνίξουν αντιγενές του. Βέβαια στην αρχή όλοι λένε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και σχέδιο Β και θα πρέπει να το διατρανώσουμε και αυτό και να πούμε ότι στην Ευρώπη αν συμφωνήσουμε μπορούμε να βάλουμε και ένα τέλος ε, ε, στην Κυριοζήνη. Υπάρχει αυτό και αλλού μπορούμε να το επιβάλλουμε ένα τέτοιο φόρο. Και με 500 εκατομμύρια κατοίκου εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπε επιβάτες, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Σικάγο, υπάρχει δυνατότητα δεν επιτρέπεται να επιβληθεί ε, φόρος στην κυροζήνη που έχει ε, στο ε, δεπόζιτό του το αεροπλάνο τη στιγμή που προσγειώνεται. Αλλά μπορείς να επιβάλλεις φόρο όταν βάζει κυροζίνη στο αεροδρόμιο ένα αεροπλάνο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γνωρίζετε και τους αριθμούς και πόσο ακριβά θα ήταν τα πράγματα. Αν δεν κινηθεί ο κόσμος, σας αρχίσουμε από την Ευρώπη. Είμαστε αρκετά ισχυροί. Αυτό που μας χρειάζεται είναι αυτοπεποίθηση. Δεν πρόκειται κανείς να πετύχει παγκόσμια ρύθμιση ε, από την προϋπόθεση ότι όλοι ε, θα πρέπει να ξεκινήσουν. Ξέρετε και το παιχνίδι με κάτω, όποιο κινηθεί πρώτο χάνει, όποιο ξυλάκι πέσει. Ε, αρχίσει η Ευρώπη, έχουμε χάσει αρκετά ω Ευρώπη. Κάποτε ήμασταν ηγέτε. Αυτά έχουν χαθεί προπολού και αν δεν κινηθεί η Ευρώπη, αν δεν κινήσει τι εξελίξει, δεν πρόκειται να κινηθεί κανένα άλλο. Αυτό να συμφωνήσουμε. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και για τον Μάτι για τα σχόλιά του. Συμφωνούμε σαφώ ε, σαφώς ε, ότι το θέμα του ανταγωνισμού συνδέεται με το σύστημα εμπορίας σταματούμε το ρολόι, αλλά δεν μπορούμε να το σταματήσουμε για όλες τις πτήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Όταν βλέπουμε πτήσεις εισερχόμενες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουν καθόλου σταματημένο το ρολόι. Ε, οι προτάσεις αυτές βεβαίως παρουσιάστηκαν πριν από μερικούς μήνες. Ε, όσον αφορά τις τροπολογίες ορισμένων συναδέλφων για τα έσοδα ε, από το σύστημα εμπορίας, αυτές τις τροπολογίες δεν θα τις υποστηρίξουμε. Εδώ μιλάμε για εταιρείε, για business εταιρείε, όχι για φιλανθρωπικές οργανώσεις και ε, αν ε, θέλαμε να ρυθμίσουμε το θέμα των εισόδων θα ήθελα να το δω να διοχετεύεται στην έρευνα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι κατάλληλο και τη στιγμής. Ανησυχώ μέχρι σε ενό βαθμού να δούμε τώρα τι θα γίνει με τη σύνοδο του ΙΚΑΟ, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξουν. Όπω είπε και η κυρία Μάισνερ, είχαμε θαυμάσει συζητήσει με του Αμερικανού φίλου μα την περασμένη εβδομάδα και ξέρετε, δεν είναι εύκολο το θέμα, καθόλου εύκολο για κανέναν. Τελικά όμω υπάρχει ακόμα το ζήτημα, ε, ένα ζήτημα με το οποίο οι Αμερικανοί συμφωνούσαν. Δεν είναι μόνο το θέμα αγορακεντρικών μέτρων ή μέτρων που στοχεύουν στην αγορά. Ε, είναι θέματα τα οποία συνάδουν ε, και με την πρόοδο της ε, έρευνας, την τεχνολογία, την ακτινοβολία και δεν είναι βεβαίως, το, τα μέτρα αυτά δεν στοχεύουν να είναι, ε, να είναι μια πανάκια η οποία θα σταματήσει και θα καταργήσει εντελώς όλων των ειδών τις εκπομπές. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει μετά το τέλος του χρόνου, αν δεν επέλθει καμία αλλαγή, διότι τότε θα πρέπει να επανέλθουμε στο πρώτο σημείο που έθιξε ο εισηγητής μας, που αφορά ανταγωνισμό, εσωτερικά δρομολόγια, εσωτερικές πτήσεις και αερομεταφορείς. Να δούμε λοιπόν τι θα, ποια θα είναι η αντίδραση της Κομισιόν. Κυρία Ντεβεράκ. Merci, Monsieur le Président. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να στηρίξω την αναβολή που μας προτείνει η Κομισιόν, που θα, πράγμα που θα καθυσυχάσει κάπως τη συζήτηση με τις τρίτες χώρες, ώστε να συζητήσουμε στο πλαίσιο της ΣΥΚΑΟ το επόμενο φθινόπωρο αυτό το θέμα. Είμαι θετική, αλλά επί της ουσίας η διαδικασία εφαρμογή αυτής της έκθεσης παραμένουν αόριστες και θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το θέμα. Για το δεύτερο εξάμεινο του 2012 μας ανακοινώνουν ότι μόνο οι ενδοευρωπαϊκές πτήσεις θα... Ε, επιβαρύνονται με, την, ε, με το, μάλλον θα συμμετέχουν στο σύστημα. Εντάξει, αλλά τότε πώς θα γίνει αυτή η αναβολή για τις τρίτες ε, χώρες. Οι ποσοστώσεις ε, ισχύουν για την μεταφορά και όχι για την αγορά. Ενώ πριν από κάποιους μήνες εμείς επιτρέπαμε στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να δέχονται μέχρι 15% πιστώσεων επί τη βάση του συνόλου των πτήσεών τους εδώ και εξοκοινωτικών. Σήμερα αλλάζουμε τους όρους επιτρέποντάς τους αυτές τις πιστώσεις να μπορούν να τι χρησιμοποιήσουν στο όριο το 15% ε, ε, ε, που αφορά τι ενδοευρωπαϊκέ πτήσεις. Θα πούμε λοιπόν σε αεροπορικέ εταιρείε που μας εμπιστεύτηκαν εμά του νομοθέτε να τους πούμε ναι, εσείς στηρίζετε τους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά ευχαριστούμε, θα αλλάξουμε τώρα ξανά του κανόνε και η ποσοστό σα είναι μια χασούρα. Ξεκάθαρη χασούρα. Και λέω ότι θα είναι χασούρι γιατί μπορούν να μπουν στην άκρη και να χρησιμοποιηθούν μέχρι το 2015, αλλά δεδομένε της μείωσης του πλαφών για την περίοδο 15-16 δεν μπορούν με το 1,5% για ένα-δύο έτη, γιατί αυτές είναι οι καλές εταιρείες που τήρησαν τις οδηγίες μέχρι στιγμής, που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα αποθέματά τους μέχρι το 2018 ε, να του πούμε τι να κάνουμε, παίξατε και χάσατε. Εμεί όμω οι νομοθέτε μπορούμε να ενεργήσουμε με τέτοιο τρόπο απέναντι σε αυτούς μα εμπιστεύονται. Γι' αυτό και προτείνω τροπολογία που δεν είναι υπέρ τη τάδε δίνα δηλαδή αεροπορική εταιρεία, αλλά που στόχο έχει να μην ε, τιμωρήσει του φορεί που τήρησαν ε, του κανόνε του παιχνίδιου και θέλω να σα ζητήσω να στηρίξετε και εσεί αυτή την τροπολογία που είναι κοινή λογική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και με συγχωρείτε που άρχισα γιατί ήμουν στην, Επιτρο... στην νομική επιτροπή. Είχαμε μια υποχρέωση εκεί. Βέβαια, από πλευρά πρασίνων, θα θέλαμε να είχαμε ακολουθήσει ακόμα πιο φιλόδοξο δρόμο, να ασκήσουμε ακόμα πιο πολύ πίεση σε αυτό τον τομέα, ε, διότι πρέπει να μην ξεχνάμε ότι όσο πιο υποχρεωτικοί είμαστε τώρα, τόσο πιο ε, πολύ θάρρο δίνουμε στους ε, αντίπαλους, ε, σε αυτούς που αντιτίθενται σε αυτό το σύστημα και θέλουν να ανατρέψουν το όλο σύστημα. Αυτή είναι η προδιάθεσή τους. Είμαι ικανοποιημένη πάντως που υπάρχει ακριβώς ε, αυτό το, έχει σημειωθεί αυτό το θέμα, ε, έχει ληφθεί υπόψη δηλαδή, ε, όχι μόνο ως μέσο οικονομικό πίεσης, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς ότι έχει δοθεί ένα σήμα να εξεταστεί η ροή αυτών των χρημάτων, αυτών των κονδυλίων, προς πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, αυτά τα ποσά. Βεβαίως θα αναγκαστώ να συμφωνήσω τρίζοντας τα δόντια μου και με μεγάλες επιφυλάξεις, αλλά τι άλλο να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος, η κυρία Μπαντίνη από την Κομισιόν. I'm sorry, that's, that's a very new pronunciation of my name. Badram, but yes. Badram λέγομαι, καμία σχέση με το πώς είπατε το όνομά μου. Κοιτάξτε, εγώ διάβασα αυτό που λέει εδώ. Βαλντίνη λέει. Ναι, ρίχτε τα στον Κρίστοφερ. λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή, καθώς και όλους όσους ε, θέλησαν να σχολιάσουν την προτινόμενη εξαίρεση. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομη και θα σχολιάσω κάποια πράγματα που υπόθηκαν. Ε, κατά Καταρχήν, είναι κάπως δύσκολο για μας από πλευράς της Κομισιόν να κατανοήσουμε τις προτάσεις για την επέκταση του πεδίου της εξαίρεσης που έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει και το, κυκλοφορία εντός ΕΟΧ. Ε, το θέμα ήταν να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην θετική δυναμική που είχε δημιουργηθεί στον ΙΚΑΟ και να δώσουμε χώρο για συζήτηση για αυτά τα θέματα, προσωρινά εξαιρώντας, ε, μάλλον αναβάλλοντας την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος ETS για την ε, κυκλοφορία εκτός πτήσεων, μάλλον εξοκοινωτικών. Ε, αν το κάναμε και για τις ενδοκινοτικές πτήσεις ε, θα ήταν κάπως αντιπαραγωγικό από τη στιγμή που προσπαθούμε να διαπραγματευτούμε ένα παγκόσμιο ETS. Τώρα όσον αφορά την Ελβετία, είναι ιδιαίτερη η κατάσταση. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για να συνδέσουμε τα συστήματα εμπορίας εκπομπών. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ελπίζουμε να έχουν αίσια έκβαση φέτος κιόλας και μάλιστα να καταλήξουν στη πλήρη σύνδεση των συστημάτων μας. Σε αυτή την περίπτωση Η Ελβετία δεν απέρριψε την ε, συμμετοχή της εξ αρχής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, οπότε Δεν θέλουμε να επεκτείνουμε την εξαίρεση και στην Ελβετία. Η Ελβετία εξάλλου έχει πολύ φιλόδοξη περιβαλλοντική ε, πολιτική και πολύ παρόμοια με αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσον αφορά την χρήση των εθνικών πιστώσεων, η εξαίρεση προτείνουμε είναι μονοετής, επειδή δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία. Η εξαίρεση, αν δεν υπάρξει μάλλον συμφωνία, η εξαίρεση θα λήξει και το ευρωπαϊκό σύστημα ETS ε θα επιβληθεί πλήρω για την ε, ε, αεροπλοεία. Δεν έχουμε δώσει εξαίρεση για κανένα άλλο κύριο τμήμα, όπως η χρήση των διεθνών πιστώσεων, αυτό εξακολουθεί να περιορίζεται στο 15% της υποχρέωσης ε, παροχής. Είναι αλήθεια ότι ορισμένοι φορείς ε, μπορεί να έχουν αγοράσει περισσότερες πιστώσεις εν ώψη μιας ε, κάλυψης 100%. Πάντοτε υπάρχει δυνατότητα να συμμορφωθεί κανείς πλήρως με το ευρωπαϊκό ETS, δηλαδή να συμμορφωθεί και με το διεθνές πεδίο ε, τρίτων χωρών. Αν κάποιος φορέας όμως θέλει να εξαιρεθεί, υπάρχουν ε, παράγοντες μείωσης στο βαθμό της οικονομικής επίπτωσης της συμμόρφωσης. Αν και δηλαδή θα τους μείνουν πελεονάσματα για τις διεθνείς πιστώσεις, εκείνα τα πλεονάσματα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια ή μπορεί να απολυθούν στην αγορά. Υπάρχει πάντοτε ένας κίνδυνος, ένα ρίσκο όταν κανείς ε, κάνει business. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι ορισμένοι φορείς έχουν περάσει το κόστος ε, της ε, συμμόρφωσης εκ των προτέρων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις υποχρεώσεις εξαίρεσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην τους μείνει το ίδιο κέρδος και αυτό δεν μπορούσε να προβλεφθεί, αλλά ζούμε σε εξαιρετικές περιστάσεις, σε προσωρινής εξαίρεσης και ελπίζουμε πως οι συνέπειες θα είναι περιορισμένο εύρος για όλους τους φορείς και ότι οι επιχειρηματικές τους αποφάσεις θα είναι δικαιολογημένες. Τώρα, τι θα γίνει μετά από την μονοετή εξαίρεση, εφόσον δεν υπάρξει κάποια συμφωνία, το, το σύστημα το ευρωπαϊκό θα τεθεί πλήρως εφαρμογή και θα ισχύει τόσο για τις διεθνείς πτήσεις όσο και για τις εσωτερικές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων μας εντός ΙΚΑΟ. Αυτά ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Μπάλτσα. Τα πρώτα τέσσερα ήταν σωστά γραμμένα, τα τελευταία τρία είχαν σοβαρές δυσκολίες. Εντάξει, γύρισαμε από τη Μεσόγειο στο Βορρά. Κυρία Φώστερ, έχετε ερώτηση? Έχω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνολική απάντηση, αλλά δεν απάντησε ακόμα στην ερώτησή μου. Κάθεστε εδώ και λέτε ε, τι θα γίνει αν στο τέλος του έτους ε, αρχίσουν όλοι να εφαρμόζουν. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είμαστε και χαζοί. Ξέρουμε τι κάνουν οι τρίτε χώρε. Ορισμένε τρίτε χώρε ήδη έχουν εγκρίνει νομοθεσία, έχουν πει στι εταιρείε του ότι σιγά μην συμμορφωθούν. Κυρία Φώστερ, ερώτηση είναι αυτό, λέει ο πρόεδρο. Μα ήθελα απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. Μπορείτε να την επαναλάβετε. Ωραία. Εσείς τι θα κάνετε τώρα, ε, Κομισιόν, αν οι τρίτες χώρες ε, εξακολουθούν στα τέλη του έτους να μην θέλουν να εφαρμόσουν, να συμμορφωθούν. Δεν ξέρω, πρόεδρε, το λέω τώρα γιατί ξεκάθαρα δεν το είπα ίσως προηγουμένως. Πολύ ξεκάθαρα το είπατε. Το θέμα αν σας απάντησαν ή όχι είναι άλλη ιστορία. Κυρία Μπάντρο μου, θέλετε να απαντήσετε. Πολύ σύντομα. Εμείς δεν έχουμε κάνει παρέκκληση ε, μόνιμη στην εφαρμογή του νόμου, προσωρινή μόνο για ένα έτος. Τελεία. I, I, I think the gist is no plan. Ε, νομίζω στην ουσία αυτό που θέλει να πει είναι ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ε, ε, λύση και σχέδιο Β δεν έχουν σκεφτεί. Ο κύριος Γκρος, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να πω το εξή για την Ελβετία. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να το αφήσουμε στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ελέγξει αν υπάρχει το νομικό πλαίσιο και για μένα αυτό μπορεί να είναι μόνο προϊόν συμφωνίας. Και θα παρακαλούσα, θα, μάλλον θα έλεγα το εξής Ας μην προεξοφλούμε από τώρα μια συμφωνία με την Ελβετία και να γράψουμε στην έκθεση ότι υποχρεούται, μα αν δεν, δεν θέλει να το κάνει, δεν πρόκειται να το ακολουθήσει αν δεν υπάρχει νομική βάση. Έτσι κι αλλιώς. Εξού και προτείνω τις τροπολογίες 22 και 13 να τις υπερψηφίσουμε, διότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται η ελόγω συμφωνία. Δεύτερον, θα ήθελα να ξαναπώ σε όλους και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Επιτροπή μας αποδίδει μεγάλη σημασία ε, στην αξιολόγηση και στην επαλήθευση, να συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Και από εκεί και πέρα να συζητηθεί μια δεύτερη φάση, το ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι, ε, που είναι τα στοιχεία που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και την αγορά, να τα λάβουμε πιο ισχυρά υπόψη και ενδεχομένως εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε και τις λεγόμενες διεθνείς πιστώσεις, διότι εναπόκειται στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο και σε εμά τα επόμενα χρόνια ε, να προσαρμόσουμε αυτό το θέμα σύμφωνα με τη διεθνή κατάσταση. Ξέρω ότι δεν είναι πολλές οι αεροπορικές εταιρείες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη δυνατότητα. Έχει δίκιο κύριε Ντεβεράκο όμως, δεν επιτρέπεται κάποιοι που έχουν ε, προετοιμαστεί να τηρήσουν μια νομοθεσία να υφίστανται κυρώσεις και κάποιοι άλλοι που ε, καιροσκόπησαν και κερδοσκόπησαν να ανταμείβονται ότι έτσι κι δεν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία. Πραγματικά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις ευλώσεις στην αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρός. Αύριο είναι η ψηφοφορία παιδιά και θα δούμε τι θα γίνει. και ποια θέση θα έχουμε. Γνωμοδότηση είναι αυτή για την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίσω το πέρα στη συνεδρίαση ε, για σήμερα. Ραντεβού στις 5 με τους συντονιστές και αύριο στην ημερήσια διάταξη με την οποία συμφωνήσατε έχουμε... Ανταλλαγή απόψεων με το Διευθυντή της ΕΑΣΑ ε, και ε, ο ίδιος ο κύριος Σκάλας θα έρθει αυτό αυτοπροσώπος να μας παρουσιάσει το τέταρτο πακέτο τη δέσμη μέτρο για τους σιδηροδρόμους και την καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές. Λοιπόν, και η Γενική Διεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σημειώστε τα αυτά. Ρεβού στις πέντε συντονιστές.